κάτι από αυτή την έκθεση το οποίο θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Δεν θα τελειώσουμε με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάλερ. Με την παρέμβασή σας ως εισηγητού κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Μια μικρή ανακοίνωση πριν περάσουμε στην επόμενη έκθεση από το ΕΛΚ Χριστιανοδημοκράτες έχω λάβει το αίτημα ορισμού ε, στην Επιτροπή για την Επιτροπή Γεωργίας συγκεκριμένα και αγροτική ανάπτυξη. Ανιές Λεμπρά, Επιτροπή Απασχόληση Κοινωνικών Θεμάτων Φιλίπ Μπουλόν, Επιτροπή Αναφορών επίση, Φιλίπ Μπουλόν. Υπάρχουν παρατηρήσεις των ορισμών αυτών. Επομένω, θεωρούνται εγκεκριμένοι. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, περνάμε στη συζήτηση τη εκθέσεω Ουγγουρεάνου, στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εύξενο πόντο. Δίνω το λόγο στον εισηγητή για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από ακριβώς τρία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την συνέργεια για τον έξινο πόντο. Ήταν ένα πρώτο βήμα προς μια πολιτική σε μια από τις πιο, σε μια από τις πιο ευαίσθητες περιοχές. Ήταν αυτό προς την κατεύθυνση, διότι ο εύξηνος πόντος αναλύεται και θεωρείται ως ένας χώρος ε, στρατηγικών ε, ελπίδων αλλά και φόβων και φιλοδοξιών. Σήμερα η πολιτική μας στον τομέα αυτό μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Το Κοινοβούλιο μπορεί να επιδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο για την αναβάθμιση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πλήρη στρατηγική. Αυτή είναι και η βασική ιδέα που διέπει την έκθεσή μου για την οποία με υποστήριξαν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και από όλο το Κοινοβούλιο. Γιατί όμω χρειάζεται νέα έκθεση για τον εύξηνο πόντο και γιατί χρειάζεται μια στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εύξηνο πόντο. Κάποιοι λένε είναι μικρή η θάλασσα αυτή. Και πράγματι είναι μικρή, αλλά αν αλλάξει ο χάρτη αυτό σε Αίγιο στρατηγικό χάρτη, τότε βλέπουμε ότι ε, προσλαμβάνει τεράστιε διαστάσει αυτή η θάλασσα. Και υπάρχει και κάτι ακόμα. Ξένο πόντο, η, η μαύρη θάλασσα όπω τη λέμε, είναι όλο και πιο μαύρη πλέον. Μετά την προσχώρηση Βουλγαρία-Ρουμανία, εν μέρη είναι μια εσωτερική θάλασσα, εσωτερική για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά οι εξελίξει στην περιοχή συχνά είναι απρόβλεπτες. Ε, υπάρχει σώρευση εντάσεων και άφθονε παρανοήσει. Αν αναλύσουμε λοιπόν την κατάσταση των ξενοπόντων θα συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν κάποιε αρνητικέ ε, προκλήσεις που όχι απλά παραμένουν αλλά και εντείνονται. Το 2008 Γεωργία-Ρωσία, ψυχρές συγκρούσεις επιδείνωση ανησυχητική του κράτους δικαίου στην Ουκρανία ή στη Ρωσία. Πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις όλες αυτές ε, που αποτελούν και ζωντανά παραδείγματα των κινδύνων ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην περιοχή αυτή. Αν εξετάσουμε τα σημερινά αποτελέσματα της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, φαίνονται μεικτά η προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον αυξημένο πόντο δεν έχει μηχανισμούς παρακολούθησης αξιολόγησης και συνέχειας. Η περιοχή αυτή δεν είναι αρκετά προβεβλημένη στις συζητήσεις ε, στις Βρυξέλλες και η κοινοτική χρηματοδότηση για την περιοχή είναι ε, κατακαιρματισμένη και πολύπλοκη θα έλεγα. Κυρία Πρόεδρε, θέλουμε να υποφεληθούμε ε, των πλεονεκτημάτων της ε, συνέργειας των πόντων η οποία εγκρίθηκε πριν από τρία χρόνια, αλλά νομίζω ότι μια νέα στρατηγική θα πρέπει να υιοθετήσει πιο στέρεες πολιτικές και συγκεκριμένα εργαλεία. Θέλω να αναφέρω δύο μόνο συστάσεις που περιλαμβάνει η έκθεσή μου. Πρώτα απ' όλα επαρκής πόρη. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διαδραματίσει ένα μείζωνα ρόλο στον ξενοπόντο θα πρέπει να το κάνει με τους απαραίτητους φόρους, πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς. Συγκεκριμένο κονδύλιο στον προπολογισμό, γιατί ο προπολογισμό είναι σημαντικός. Δεύτερον, εκπόνηση ενό σχεδίου δράση Ευρωπαϊκή Ένωση με σαφεί στόχου, σαφή καθήκοντα. Μεταξύ αυτών, τακτέ συναντήσει σε υπουργικό επίπεδο των χώρων της ε, περιοχής η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ΑΕΦ πόντων δεν θα πρέπει ούτε να υποτιμά αλλά ούτε και να υπερεκτιμά οποιοδήποτε από τα κράτη της περιοχής. Η αρχή της ε, αλληλεγγύης, ε, της ε, εταιρική σχέση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας ό,τι αφορά την περιφερειακή συνεργασία, αλλά και όλους τους άλλους περιφερειακούς εταίρους. Για να ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την πολύ θετική συμβολή τους στην τελική έκδοση της, εκδοχή της έκθεσής μου και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι το Κοινοβούλιο αυτό το οποίο αναμένει και από το Συμβούλιο αλλά και από, το, και από την Κομισιόν είναι να δώσει σάρκα και οστά στην έκθεση αυτή για μια στρατηγική συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή του έξουν πόντου. Να αποτελέσει αυτό μια πραγματικότητα. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Σικτά. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φίλεξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι η Μαύρη Θάλασσα είναι σοβαρό θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σημαντική περιοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να εστιάσουμε εκεί για να δείξουμε πως έχει μεγάλη ευαισθησία για μας. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή, τον κύριο Τραϊάν Ογκουρεάνου και την Επιτροπή Εξωτερικών για μια ουσιαστική και εξαιρετική έκθεση. Οι συστάσεις είναι ενδιαφέρουσες και καινοτόμες σε πολλά ζητήματα. Από την τελευταία διεύρυνση η Μαύρη Θάλασσα είναι και ευρωπαϊκή θάλασσα. Έχουμε λοιπόν κάποιες ευθύνες ε, όπως έχουμε και έναντι όλων των άλλων λεκανών που βρέχουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την ευθύνη. Ως μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας έχουμε ήδη ένα στόχο πρωτοβουλία τη συνέργεια δηλαδή της Μαύρης Θάλασσας. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε πως η εφαρμογή έχει αποδειχθεί πολύ πιο δύσκολη από όσο αρχικά νομίζαμε δεν καλωσορίζονται όλοι οι στόχοι μας με ενθουσιασμό από όλους στην περιοχή. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο το Κοινοβούλιο έχει επιλέξει μια προσέγγιση που βασίζεται στο ότι θα πρέπει να το νιώθουν δικό τους αυτό οι χώρες περιοχής και βεβαίως την ενίσχυση του διαλόγου. Είναι σωστή αυτή η προσέγγιση. Αλλά οι δεσμεύσεις αυτές μπορούν να είναι αξιόπιστες εάν και όταν ε, αποδεικνύονται ουσιαστικές βελτιώσεις στην ζωή των πολιτών και άρα έτσι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μία νέα ευρωπαϊκή στρατηγική η οποία θα αντιπροσωπεύει την δέσμευσή μας για την περιοχή και για τα κράτη-μέλη που ανήκουν στην περιοχή αυτή δίνοντας την πλήρη στήριξή μας για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την γεωγραφική τους κατάσταση. Αντιλαμβανόμαστε πως η στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να ερμηνευτεί ως ε, αντικατάσταση των υπαρξιών προσπαθειών, όπως παραδείγματο χάρη της συνέργεια για τη Μαύρη Θάλασσα. Πρέπει να είναι ένα συνολικό πλαίσιο που μπορούμε να δώσουμε κατευθύνσεις για όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης στην περιοχή. Η στρατηγική της Μαύρης Θάλασσας μπορεί να αποτελέσει ιδανικό βήμα για να ανανεώσουμε το ενδιαφέρον μας στην περιοχή και μιλάω εδώ πέρα για τα στρατηγικά, πολιτικά και οικονομικά συμφέροντά μας και να δούμε πώς μπορούν να επιτευχθούν. Το Κοινοβούλιο έχει δει τα βασικά πεδία στα οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η στρατηγική, δηλαδή διακυβέρνηση, ασφάλεια, ενέργεια, μεταφορές περιβάλλον και βεβαίως ε, εμπόριο και οικονομική ανάπτυξη και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Αυτή η στρατηγική βεβαίως μπορεί να προσθέσει μια θαλάσσια διάσταση στις δραστηριότητες μας και αυτή τη στιγμή η Κομισιόν αναπτύσσει ένα συνολικό πακέτο που θα αναφερθεί στις πρωτοβουλίες θαλάσσιας πολιτικής, διαχείρισης των φυσικών πόρων και ε, βεβαίως ε, καταπολέμηση της ελαφραλίας μπορούμε εδώ πέρα να αντλήσουμε εμπειρία από άλλες στρατηγικές όπως τη στρατηγική για τη Βαλτική και τη στρατηγική για τον Δούναβη. Η δε στρατηγική για τον Δούναβη προφανώς θα έχει αλληλεπίδραση με τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά γνωρίζουμε πως κάθε ευρωπαϊκή λεκάνη είναι διαφορετική. Οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε πως όλες οι μελλοντικές ευρωπαϊκές στρατηγικές ε, θα προσαρμοστούν στα τομιακά τους χαρακτηριστικά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, των περιβάλλον, την ενέργεια, υποδομές και φυσικούς πόρους. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η έκθεση για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής της Ένωσης για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας προσφέρει μια γενική εικόνα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή αλλά θα πρέπει να αναπτύξουμε και σταθερούς διάβλους με τις χώρες περιοχής για να υπάρχει ομαλή εφαρμογή. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να έχουμε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους, ξεκινώντας με τους εταίρους μας ε, στην περιοχή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε καλωσορίζουμε αυτή την έκθεση και θέλουμε να αντλήσουμε από τα συμπεράσματα της Υπηρεσίας Κομισιών και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα δεσμευτούν για να προετοιμάσουν μια στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα και βεβαίω θα ζητήσουμε τη στήριξη δική σας και του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Τρεις παρεμβάσεις από ένα λεπτό, το τονίζω, από τις αρμόδιες επιτροπές με πρώτο τον κύριο Καζάκ από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, συγχαίρω τον κύριο, τον κύριο Ουγγουρεάνου που είναι ο συντάκτης έκθεσης. Ως υπεύθυνο της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ χαίρομαι που οι προτάσεις μας ελήφθησαν υπόψη. Μετά την ε, ένταξη της Βουλγαρίας και της ε, Ρουμανίας το 2007 η Μαύρη Θάλασσα έγινε Ευρωπαϊκή Θάλασσα και χρειάζεται πλήρη ευρωπαϊκή στρατηγική. Αυτό σημαίνει και διοικητικού και ανθρώπινου και οικονομικού πόρου και καλύτερο συντονισμό και λογοδοσία. Θα πρέπει η νέα στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα να βασίζεται σε συγκεκριμένα προγράμματα. Θα πρέπει να δούμε το περιβάλλον, τι μεταφορέ, τις, α, ε, ε, τους φυσικούς πόρους α, ε, σημαντικοί για την ανάπτυξη της περιοχής. Θέλουμε επίσης έντονη συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και διμερή συνεργασία, αλλά και με την κοινοβουλευτική συνέλευση του Οργανισμού Παρευξήνια συνεργασία και την Οικονομική Συνεργασία στον Εύξηνο Πόντο. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη της περιφερειακές πρωτοβουλίες. Ε, διακόπτεται ο μιλητής. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή Έρευνας και Βιομηχανίας ε, συμφωνεί με το ρυθμιστικό πλαίσιο και ενθαρρύνει τα κράτη της ε, περιοχής ε, της Μαύρης Θάλασσας να επικυρώσουν τη συνθήκη για την ενέργεια, για τη χάρτη της ενέργειας. Επίσης η Τράπεζα Ανάπτυξης και Επενδύσεων βοηθάει πάρα πολύ την περιοχή. τονίζουμε τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας. προγράμματα όπως το Ναμπούκο πρέπει να είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επίσης, ο πανευρωπαϊκός ε, ε, πέτρελαγωγός είναι σημαντικές δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαύρη Θάλασσα, όπως και η συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής. Νομίζουμε ότι αν υπάρξει ένα δίκτυο έρευνας και συνεργασίας είναι πολύ σημαντικό και καλούμε την Κομισιόν να υποστηρίξει τα προγράμματα έρευνα στην περιοχή. Ζητάμε τέλος από την Κομισιόν να εφαρμόσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή με ένα σχέδιο δράσης και χρειάζεται ε, υπάρχει, να υπάρξει και ένα σύνδεσμος με τη στρατηγική ε, για την περιοχή του Δούναβη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποστινάρου ε, από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η σημασία της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις για τις μεταφορές, για την ενέργεια, για το περιβάλλον και για τη σταθερότητα της περιοχής είναι σημαντική. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή θα έχει θετική επίπτωση στην περιοχή αυτή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το συνόλο της. Η Επιτροπή μας πιστεύει ότι θα μπορούσε η στρατηγική μας να οδηγήσει σε βιώσιμη ε, ανάπτυξη ε, για την περιοχή. Όμως, για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει όλα τα κράτη της περιοχής να εμπλακούν, είτε ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε όχι. Αυτή η στρατηγική χρειάζεται συντονισμό στις δράσεις της και πώς θα μπορούσε να υπάρξει αυτός ο συντονισμός χωρίς να εμπλακούν όλες οι χώρες. Ο συντονισμός χρειάζεται όμως και με τη στρατηγική για το Δούναβη που υποτίθεται ότι θα γίνει μεγάλη προτεραιότητα της Ουγγρικής ε, Προεδρίας. Το να υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση και διαπεριφερειακή συνεργασία θα πρέπει να υπάρχει σε όλους τους τομείς, αλλά κυρίως στην ενέργεια, στις μεταφορές και στο περιβάλλον. Ευχαριστώ τον κύριο Ποστινάρου. Τώρα, ο κύριος Μπροκ από τις ομάδες. Ε, για δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει και έχει συμβάσει πάρα πολλές σκέψεις εδώ πέρα για να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Δεν πρέπει βεβαίως να μπερδέψουμε τη συνεργασία αυτή με την ανατολική εταιρική σχέση ούτε βεβαίως με τις στρατηγικές μας σχέσεις με τη Ρωσία και την Τουρκία. Είναι διαφορετικά πράγματα, αλλά από την άλλη βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι μπορούμε να συνδέσουμε όλα αυτά τα πράγματα και να έχουμε μια συνεκτική πολιτική που θα είναι προς το συμφέρον μας, θα βοηθήσει τις χώρας και να βοηθήσει στο να συμβιβαστούν αντίθετα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα και έτσι να αποφευχθούν στο μέλλον αντιπαραθέσεις ή να είναι λιγότερο επικίνδυνες και δραματικές όπως παραδείγματο χάρη με την ανατολική μας εταιρική σχέση η οποία δεν είναι εναντίον κάποιου παραδείγματο χάρη βλέπετε πως οι ευρωπαϊκές ε, προοπτικές έχουν ε, διαφορετική μορφή από ό,τι παραδείγματος χάρη ε, με την Ρωσία. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν αυτή η διάκριση, κάτι το οποίο οπωσδήποτε ξέρει ο κύριος Επίτροπος, αλλά νομίζω πως γι' αυτό το λόγο η συνεργασία της Μαύρης Θάλασσας είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ρωσίας, της Τουρκίας και των υπολείπων χωρών που ανήκουν στην ανατολική εταιρική σχέση. Και φαντάζομαι πως ε, θα συνεισφέρει αυτό στις ε, καλές σχέσεις με τις χώρες περιοχής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπρόκ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος Πάσκου για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εύξενος πόντος είναι μία πύλη προς και από την Ευρώπη και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι ένα μακρινό, απόμακρο μέρος του κόσμου το οποίο προσελκύει που και που την προσοχή μας υπάρχουν θέματα σε μερίσια διάταξη τα οποία έχουν να κάνουν με την παρευξήνια περιοχή όπως διακοπή της διακοπής φυσικού αερίου 6-8 ή ο Γεωργιανός πόλεμος το 2008. Παρά όμως τις αποδείξεις και τα στοιχεία που έχουμε η παρευξήνια περιοχή δεν έχει ακόμη την περιοχή που της αρμόζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν υποχρεώθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά όταν προσχώρησαν στην Ένωση Ρουμανία και Βουλγαρία το 2007. Η συνέργεια των πόντων οποία εκπονήθηκε με, λίγο μετά την προσχώρηση των δύο χωρών, αναδρομικά φαίνεται ότι ήταν μια βεβαιασμένη κίνηση, ένα έγγραφο ε, το οποίο θέλησε να καλύψει αυτό το λευκό σημείο ή αυτή τη μαύρη τρύπα, ανάλογα με το πώς θέλετε να το πούμε, σε αυτό στο χάρτη. Αλλά σε ό,τι αφορά την πρώτη αναθεώρηση που έπρεπε να γίνει το 2008, δεν είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα, ούτε και η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής, της συνέργειας αυτής ε, είναι πολύ αισιόδοξη. Θέλω να πω ότι φαίνεται να μην υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά και φαίνεται να υπάρχει και απροθυμία να αντιμετωπίσουν οι εταίροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν την περιοχή, ιδίω όταν υπάρχει έλλειψη χρημάτων. Αυτή η απροθυμία αυξάνεται. Επίσης η αρχική υπόθεση στην οποία βασίστηκε η συνέργεια, δηλαδή ότι η περιοχή θα πρέπει να γίνει μια περιοχή συνεργασίας που θα πρέπει να προσελκύει την προσοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την ε, στήριξη έχει αγνοήσει την αλήθεια ότι είναι τελείως διαφορετική η περιοχή αυτή από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Πώς θέλουμε να είναι συνεκτική αυτή η περιοχή και να αποκτήσει μια συλλογική ταυτότητα. Αυτό είναι ανεδαφικό για να μην πω ότι είναι και κακοπροαίρετο τώρα, σε ό,τι αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Ευχαριστώ και ως Βάλ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η έκθεση που ετοίμασε ο συνάδελφος Ουγγουρεάνου είναι πολύ ενδιαφέρουσα, τον ευχαριστώ και στρέφει την προσοχή μας ξανά σε αυτή την περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια ποικιλομορφία ε, πολιτικών συστημάτων, θρησκειών, ε, πολιτιστικών ε, κληρονομιών. Υπάρχουν διαφορές και στους φυσικούς πόρους. Υπάρχουν πολλές διαφορές. Επίσης η κατάσταση είναι τώρα είναι νέα και διαφορετική και οφείλεται στο γεγονός ότι τώρα υπάρχουν τρεις ε, χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή. Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι πολύ σημαντική για τη γεωστρατηγική της θέση που αποτελεί μια προστιθέμενη αξία και παράλληλα αλλά δημιουργεί και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια. Θα ήθελα να μιλήσω για την ενεργειακή ασφάλεια σε αυτό το επίπεδο. Το να εξασφαλίσουμε ε, σταθερή ενεργειακή παροχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης πρέπει να επηρεάσουμε στα εκρεμή ζητήματα ε, που υπάρχουν ακόμα για την περιοχή και να επηρεάσουμε και τη συνεργασία και τη σχέση μας με τη Ρωσία. Ε, θα πρέπει να συνεργαστούν όλες οι, χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες, να υπάρξει συνεργασία με τους άλλους περιφερειακούς οργανισμούς και να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Μην ξεχνάμε και την ε, τις κοινωνίες των πολιτών με τις οποίες ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε. Θα υπάρξουν και νέοι φορείς, ε, χρειάζονται αυτοί για να υπάρξει ε, τακτική χρηματοδότηση και μεγαλύτερη πολιτική εμπλοκή. Κύριε Επίτροπε, ελπίζω να χρησιμοποιήσετε αυτή την έκθεση. Ο κύριος Βέρνερ Σούλτς, για ένα μισή λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, για να γίνει η Μαύρη Θάλασσα ένας χώρος ε, σταθερότητας, ασφάλειας, δημοκρατίας και ευημερία και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Το ψήφισμα αυτό το επιτυγχάνει, γι' αυτό και το στηρίζει η ομάδα μας. Βεβαίως υπάρχουν και διάφορες άλλες προτάσεις εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη το τι θα γίνουν οι άλλοι συγκρούσεις στην περιοχή, το τι θα γίνει με την κοινωνία των πολιτών, τα έργα people to people και η στήριξή τους και η στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διασυνοριακή συνεργασίας. Επιπλέον θέλουμε μια αηφόρο ενεργειακή πολιτική, μεγαλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα και βεβαίω δημιουργία ακαδημαϊκών και φοιτητικών δικτύων. Αυτό το οποίο λείπει είναι πως δεν υπάρχει μια ενιαία στάση όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές. Ε, αναφέρομαι εδώ πέρα στον Αμπούκο και το South Stream και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ζητάμε καλύτερη επιτήρηση, ε, γιατί μάλλον αυτό το οποίο ζητήσαμε εμείς, δηλαδή καλή επιτήρηση των πλατφορμών άντλησης πετρελαίου μετά την καταστροφή του Μεξικού δεν γίνεται δεκτό. Θα ξανακαταθέσουμε την ε, τροπολογία. Ευχαριστώ. Κύριο Σκόβαλ για ένα λεπτό. E, Κυρίες και κύριοι, κύριε Πίτροπε, το έγγραφο που έχει συνταχθεί αξίζει της υποστήριξής μας. Εκ μέρους της ομάδας μου εκφράζω αυτήν την υποστήριξη. Η συνέργεια για την ε, Μαύρη Θάλασσα θα πρέπει να επανεξεταστεί γιατί ορισμένες καλές ιδέες δεν έχουν μεταφραστεί σε πρακτικές ε, δράσεις. Το βασικό καθήκον του κυρίου Φιουλε θα πρέπει να είναι να βάλει τάξη σε αυτή την ευρωπαϊκή περιοχή και να δείξει ότι η πιο σημαντική από τις πολιτικές γειτονίας μας ε, προσθέτει κάτι στην περιοχή. Χρειαζόμαστε σταθερότητα ε, σε, αυτό το, σε αυτή την περιοχή ε, και σταθερότητα και στον τομέα της ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο που υποστηρίξουμε και τη γεωργία στην ε, μεταρρυθμιστική της προσπάθεια. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτή την προσπάθεια, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι και αποτελεσματική. Κάμπελ Μπάνερμαν, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, όταν μιλάμε για τη Μαύρη Θάλασσα, μία λέξη μας έρχεται κατά νου. Προσοχή. Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η Μαύρη Θάλασσα είναι η αυλή της ε, Ρωσίας, έχει ναύσταθμο στην ε, Κρυμαία, σεβαστό πολύ κοντά στα πεδία μαχών του Δευτέρου Παγκοσμίου. Είδαμε τι έγινε στην Γεωργία. Εάν η Γεωργία ήταν στο ΝΑΤΟ, οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές. Αν και υποστηρίζω την ανεξαρτησία της Γεωργίας, δεν είναι σωστό να προκαλεί κανείς τη ρωσική αρκούδα στη φωλιά της. Μετά υπάρχει η Τουρκία, με την οποία παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της προσφέρει ένταξη παρά το ότι μέλη όπως η Γαλλία θα ασκήσουν βέτο. Η Τουρκία έχει 4% της έκτασης της στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι στο να παραπλανούμε την Τουρκία. Η απογοήτευση θα μπορούσε να οδηγήσει την Τουρκία στα χέρια Ισλαμιστών εξτρεμιστών. Και βεβαίως ε, μην ξεχνάμε πως η Μαύρη Θάλασσα περιέχει πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ευχαριστούμε λοιπόν τον κύριο. Τον λόγο έχει ο κύριο Στογιάννοφ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, προσυπογράφω σε πολλές από τις απόψεις ε, που ακούστηκαν και θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Από την αρχαιότητα περιοχή αυτή είχε οικονομική και πολιτική σημασία για την Ευρώπη και συνεχίζει να έχει την ίδια σημασία μέχρι σήμερα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η στρατηγική. Η ίδια συζήτηση επαναλήφθηκε πρόσφατα. Θα ήθελα τώρα να τονίσω κάτι το οποίο αναφέρθηκε από τους σοσιαλιστές Θέλω να στηρίξω την πρόταση για την ε, καθιέρωση μιας ξεχωριστής γραμμής στον προπολογισμό και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περάσει στα έργα, να μεταφράσει τα όσα ακούγονται σήμερα στο ημικύκλιο σε πράξεις, που είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Γκουρεάνου για την πρωτοβουλία του σε ό,τι αφορά δηλαδή την έκθεση αυτή την οποία εκπώνησε για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εύξηνο πόντο. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που προηγήθηκαν εμού και είπαν ε, ότι πρέπει να έχουμε αυτή την στρατηγική. Η θάλασσα είναι η εστερική θάλασσα της Ευρωπαϊκή Ένωση, Έχει γεωστρατηγική σημασία που κανείς δεν μπορεί πιστεύω να την υποτιμήσει δεδομένης περιφερειακής σταθερότητας, της διαδικασίας εκδημοκρατισμού, της αναεριακής ασφάλειας και των εμπορικών ζητημάτων που ενέχονται. Νομίζω ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επωφεληθούμε και από τις δυνατότητες ε, της ε, παρευξήνιας περιοχής. Για να πετύχουμε το στόχο αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βασίζεται περισσότερο ε, στις παρευξήνιες χώρες που είναι μέλη της και θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερο δυναμισμό ηγεσία και όραμα σε σχέση με το παρελθόν. Χωρίς να επισέλθω στα ζητήματα που έχουν να κάνουν τη διαδικασία της διεύρυνσης, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όλους όσους είναι σκεπτικιστές στην παρεξήνια περιοχή. Οποιαδήποτε επιβράδυνση της διαδικασίας ε, θα ε, φέρει πίσω και τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της ε, περιοχής. Διακυβεύεται η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Οι επιπτώσεις της αστάθειας θα ήταν πολύ δύσκολο να προβλεφθούν κατακλείδη κύριοι συνάδελφοι, χρειάζεται την εσωτερική της Ευρωπαϊκή Θάλασσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την περιφέρεια και τη στρατηγική αυτή θα πρέπει να την εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των συστάσεων του εισηγητή μας. Και βέβαια το Κοινοβούλιο θα πρέπει σήμερα να στηρίξει με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίγκλερ. Κυρία Κοπά για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε σήμερα μια πολύ σημαντική έκθεση σχετικά με μια ιδιαίτερη περιοχή κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Εύξηνο Πόντο. Η περιοχή συνδυάζει χώρε τη Ένωση αλλά και χώρε σημαντικέ για την περιφερειακή συνεργασία. Είναι λοιπόν κοινή ανάγκη να διασφαλιστεί η ύπαρξη ενό χώρου ειρήνη, δημοκρατία, ασφάλεια και σταθερότητα γύρω από τον Εύξηνο Πόντο έχουμε ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας μέσα από τη συνέργεια για τον εύξεινο πόντο που έχει δρομολογηθεί εδώ και καιρό όχι όμως με απτά αποτελέσματα. η επιτυχή υλοποίησή της με τη δραστηριοποίηση όλων των χωρών που συμμετέχουν θα ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση μας στη βάση των κοινών αξιών. πρέπει δε να δράσει συμπληρωματικά με την εδρεωμένη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και την ανατολική εταιρική σχέση. η σταθερότητα και η ασφάλεια του εύξεινου πόντου έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευρώπη συνεπώς η ευρωπαϊκή ένωση μοιράζεται την ευθύνη για τη στήριξη της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. η περιοχή αυτή έχει σημασία για την ένωση ιδιαίτερα λόγω των συνδέσεων ενέργειας και μεταφορών που διαθέτει. η ενίσχυση της δημοκρατίας και ένα ισχυρότερο σύστημα κράτους δικαίου θα διευκολύνουν το εμπόριο τις επενδύσεις και την κινητικότητα των προσώπων. συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη να καταρτιστεί ειδική γραμμή του προπολογισμού για τη συνέργεια του εύξεινου πόντου αυτό θα βοηθήσει αποτελεσματικά στον εξυγχρονισμό της περιοχής. είναι στο χέρι μας κυρία πρόεδρε με τις πολιτικές μας να φέρουμε αυτές τις χώρες ακόμα πιο κοντά στην ευρώπη για το αμοιβαίο καλό όλο. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Κυρία Βαλέαν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, από το 2007 Αναγνωρίσαμε τη σημασία της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας, όμως η επίπτωση της προσέγγισής μας ήταν πολύ μικρή. Κανένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, κανένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική δράση, ένα σχέδιο δράσης ε, με προτεραιότητες, με ορόσημα, καλύτερο ε, διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών θα πρέπει ε, η εταιρική σχέση για την ενέργεια και τις μεταφορές ε, να ε, υπάρξει, μαζί με την εταιρική σχέση για το περιβάλλον. μόνο με μικρά, μικρής εμβέλειας προγράμματα μπορούμε να έχουμε σημασία. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε την κατακαιρματισμένη προσέγγισή μας και για τα οικονομικά. Μέχρι στιγμής είχαμε διάφορα οικονομικά εργαλεία, αλλά δεν είχαν ουσιαστική επίπτωση. Γι' αυτό η το κοινό πρόγραμμα για τη Μαύρη Θάλασσα θα πρέπει να είναι το βασικό εργαλείο για τη στρατηγική για την Μαύρη Θάλασσα και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να προσελκύσουμε επενδύσεις και να προωθήσουμε τη συνεργασία. Ο κύριος Βλάζακ για ένα λεπτό. Ναι, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι. Η αργή εφαρμογή των προγραμμάτων, η έλλειψη σχεδίων δράσης και εκθέσεων αξιολόγησης και η έλλειψη συναντήσεων υψηλού επίπεδου και η κίνδυνη με την ανατολική εταιρική σχέση δείχνουν πως η απόφαση να πάει η ευθύνη στα κράτη-μέλη δεν ήταν η ορθότερη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παίξει μεγαλύτερο ρόλο ως γραμματεία για να διευκολύνει τη στρατηγική της Μαύρης Θάλασσας. Επίσης θεωρώ πως η στρατηγική πρέπει να προσθεθεί με τις άλλες μακροπεριφερειακές στρατηγικές και να πάει σε ένα και να είναι ουδέτερη από θεσμικής και ε, δημοσιονομικής πλευράς. Δεν θα πρέπει να έχουμε περαιτέρω πόρους ή νέα νομοθεσία ή νέα γραμματεία. Δεν χρειαζόμαστε άλλες γραμμές του προϋπολογισμού. Χρειάζεται να εστιάσουμε στην εφαρμογή συγκεκριμένων έργων που θα είναι προς συμφέρον μας. Ο κύριος Κουμουτσάκος, Πρόεδρε. 1,5 λεπτό. Είναι κοινοτυπία πλέον να υπογραμμίζει κανείς ότι η Μαύρη Θάλασσα είναι περιοχή στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, αφού μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας είναι σχεδόν εσωτερική θάλασσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενέργεια, ασφάλεια, σταθερότητα και βέβαια δημοκρατία είναι τομείς εχμής του ενδιαφέροντός μας για αυτή την περιοχή. Από το 2007 όταν ξεκινήσαμε την πολιτική μας σε αυτή την πολλαπλά κρίσιμη περιοχή έως σήμερα είχαμε ορισμένα βήματα προόδου και ορισμένες επιτυχίες. είχαμε όμως δυστυχώς και καθυστερήσεις και αποσπασματικές προσεγγίσεις και περιόδους αδράνειας. είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι από το 2008 δεν έχει οργανωθεί οποιαδήποτε υπουργική συνάντηση για την πολιτική αυτή. αυτή η κατάσταση υπολείπεται των αρχικών φιλοδοξιών μας και με δεδομένη την γεωστρατηγική γεωπολιτική και οικονομική σημασία της περιοχής δεν έχουμε παρά μία επιλογή την ενίσχυση τη πολιτική και των δράσεών μα στον εύξηνο πόντο στη μαύρη θάλασσα. υποστηρίζω λοιπόν ανεπιφύλακτα την προτινόμενη από τον εισηγητή κ. γκουρεάνο αναβάθμιση τη Ευρωπαϊκή Πολιτική για την μαύρη θάλασσα σε ολοκληρωμένη στρατηγική που θα υποστηρίζεται από χωριστή δική τη γραμμή προπολογισμού. στο πλαίσιο αυτό θέλω να τονίσω και ω μέλο τη Επιτροπή μεταφορών και τουρισμού την σπουδαιότητα αυτών των δύο τομέων που θα πρέπει απαραίτητα να είναι συστατικά στοιχεία μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη μαύρη θάλασσα. Τέλο, είναι περιττό να υπογραμμίσω ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης μπορεί και εκείνη να συμβάλει ουσιαστικά στην ενιαία βιώσιμη ανάπτυξη τη περιοχή του ευξήνου πόντου. αυτά θα πρέπει να γίνουν τώρα. Όμω η διεύρυνση είναι άλλο ζήτημα που χρειάζεται πολλή μελέτη και πολλή προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Κυρίλοβ για 1,5 λεπτό. Με την ένταξη της Βουλγαρίας και Ρουμανίας, η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έγινε όμορη περιοχή της Ευρώπης. Είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, ε, της Κασπίας και της ε, Κεντρικής Ασίας. Η γεωπολιτική και η οικονομική ε, σημασία αυξάνει σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ενέργεια. Η Ένωση θα πρέπει να αυξήσει την παρουσία της, να έχει ενεργές πολιτικές και να βρει μακρόπνοε λύσεις στα προβλήματα της περιοχή. Όλες οι παράκτιες περιοχές δεν δείχνουν ε, ενδιαφέρον για την ε, συνεργασία. Όμως αυτή είναι πολύ σημαντική ε, για να ξεπεραστούν οι συγκρούσεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε τα θέματα που μας ανησυχούν και που ενδιαφέρουν όλες τις παράκτιες περιοχές θαλάσσια ασφάλεια τα πρόσφατα χρόνια αυξάνονται τα ατυχήματα με απώλεια ανθρωπίνων ζώων και περιβαλλοντικές ζημιές στη Μαύρη Θάλασσα. Ε, θα πρέπει να μειώσουμε τα ατυχήματα αυτά βοηθώντας στις επιχειρήσεις διάσωσης στα πλαίσια της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής. Σύντομα θα ε, ασχοληθούμε με την έκθεση αυτή που ασχολείται ε, για πρώτη φορά με αυτές τις πολιτικές στη Μαύρη Θάλασσα. Ε, είναι καλή βάση και για την πολυμερή συνεργασία στην περιοχή. Ε, επίσης υπάρχουν προγραμμάτα, προγράμματα όπως ο διάδρομος, ο πανευρωπαϊκός διάδρομος 8 και 9. Ε, θέλω να ευχαριστήσω το συνάδελφο που συνέταξε αυτή την ε, έκθεση ο κύριος Σίβη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για την περιοχή του έξινου πόντου πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος τόσο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι ένας χώρος τόσο αντικρουόμενων συμφερόντων και διανέξεων επίσης. Νομίζω ότι θα πρέπει να πούμε ότι ε, δεν ε, είναι ένα ευχολόγιο αυτό, ούτε μπορούμε να λύσουμε εμείς όλα τα προβλήματα, όπως τα ενεργειακά, παραδείγματο χάρη, όταν ε, αντιτίθεται η Ρωσία στις δικές μας προτάσεις. Ούτε μπορούμε να επιλύσουμε όλες τις συγκρούσεις. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Όταν μιλάμε για την συνέργεια για τον εύξηνο πόντο είναι μια προσθέμενη αξία και πρέπει να διαρωτηθούμε γιατί δεν συνεργάζεται με άλλες περιφερειακές οργανώσεις ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι η κοινοβουλευτική συνέλευση του ευξήνου πόντου για παράδειγμα. Αυτοί θέλουν να συνεργαστούν μαζί μα, αλλά από ό,τι φαίνεται εμεί ε, θεωρούμε ότι είμαστε πολύ σημαντικοί για να ασχοληθούμε με την συνεργασία αυτή. Νομίζω όμω ότι πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Ο κύριο Κούτα για ένα λεπτό τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η περιοχή αυτή έχει μια στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υπήρχε διαθροτική στρατηγική, δεν υπήρχε σχέδιο δράσεως για την συνέργεια στη Μαύρη Θάλασσα και η χρηματοδότηση γίνεται, γίνεται μέσα από ασυντόνιστα ε, μέσα και εργαλεία. Γι' αυτό χρειάζεται μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μαύρη Θάλασσα με τον ίδιο βαθμό προτεραιότητας με τις υπόλοιπες περιφερειακές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, με βάση την οικονομική, κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη, σημασία στο περιβάλλον και στις μεταφορές και καλή διακυβέρνηση. Υπάρχουν ε, βασικά προγράμματα, ε, ο αγωγός Ναμπούκο που θα βελτιώσει την ενεργειακή μας ανεξαρτησία, η δημιουργία και ανάπτυξη λιμένων στην Μαύρη Θάλασσα. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν μόνο στα πλαίσια μιας κοινή στρατηγικής. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο Catch the Eye. Πρέπει να κάνω μια διαλογή, δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε όλους. Καταρχήν, η κυρία Σαβέλα, για ένα λεπτό έχει το λόγο. θάλασσας είναι πάρα πολύ σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Ε, κυρία Πρόεδρος, κύριε Επίτροπε, υπάρχει το μεγάλο θέμα του Ναμπούκο, από το οποίο εξαρτάται ένα μεγάλο μέρος της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Ό,τι όμως αφορά τον προμηθευτή του μεγάλου αυτού αγωγού είναι πάρα πολύ ασαφές. Χθες ο πρόεδρος της επιτροπής ο κύριος μπαρόσο μας είπε ότι ήταν στο αζερμπαϊτζάν στο τουρκμενιστάν και ότι πήγε πάρα πολύ καλά. τι σημαίνει αυτό; θα πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε ένα χρονικό όριο πότε ξέρουμε ότι είναι βιώσιμος ο ναμπούκο ή όχι να μην σπαταλάμε δυνάμεις και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε το θέμα λοιπόν του ναμπούκο το οποίο είναι από τα κυριότερα θέματα στην ενεργειακή ασφάλεια της ευρώπης είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ξεκαθαρίσει έχουμε προμηθευτεί ή όχι. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. σας ευχαριστώ. θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο λουάν για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκουρεάν για την εξαιρετική του έκθεση. Μια έκθεση πάρα πολύ σημαντική και από γεωπολιτική όσο και πολιτικής πλευράς, οικονομικής πλευράς. Είναι πολύ μεγάλο το δυναμικό της περιοχής και στον τομέα της ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν να προβληθεί και το θέμα της ασφάλειας ε, του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενέργειε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, έχουν γίνει, δεν ήταν ιδιαίτερα ξεκάθαρε και η συνέργεια για τον εύξενο, πόντο δεν είχε τα προεξοφληθέντα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ΕΙΕΔ, ελπίζω να έχει απαραίτητου πόρου ε, και ανθρώπινου και χρηματοοικονομικού για να εφαρμόσει τις ε, τρει εταιρικέ σχέσει δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε την περιοχή αυτή. Θα πρέπει να σηματοδοτήσουμε την παρουσία μας εκεί με συνεκτικές δράσεις, μακρόπνες δράσεις που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της, χώρα, της περιοχής αυτής. Ζέγγιντι, ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ως βουλευτής πρέπει και εγώ να πω κάποια πράγματα γιατί επί Ουγγρικής Προεδρίας υπάρχει κάποια σχέση με την ε, στρατηγική αυτή. Υπάρχει λοιπόν ένα περιφερειακό σχέδιο ανάπτυξης και η στρατηγική του Δούναβη μπορεί να είναι αξιόπιστη μόνο αν είναι ανοιχτή και προς άλλες περιφερειακές ε, στρατηγικές. Και δεύτερον, η ενεργειακή ασφάλεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εάν θέλουμε να αποκαταστήσουμε την ειρήνη στην ε, περιοχή, τότε πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε συγκεκριμένα βήματα στην περιοχή για την ενεργειακή ασφάλεια. Όπως ξέρετε και ακούσατε χτες η ενέργεια είναι βασική προτεραιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βανίστελ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Μαύρη Θάλασσα είναι πάρα πολύ κοντά μας, είναι Ευρωπαϊκή Θάλασσα και αν δούμε και την ε, ε, οπτική γωνία της ε, ενέργειας καθώς είμαι και σκιοσηγητής για το ΕΛΚ έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές εκεί πέρα και βέβαια το κλειδί είναι η συνεργασία μιλήσαμε για ε επενδύση στον Αμπούκο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με σταθερέ σχέσει. Ο Μπαρόσο είπε χθε πώ είχε αποτελέσματα στο Αζερβαϊτζάν και το Τουρκμενιστάν. Δηλαδή η προστιθέμενη αξία είναι σαφής και νομίζω τα ανέφερε και ο κύριος Μπροκ. Οπότε το να έχουμε πολλές πηγές ενέργειας είναι κατά την άποψή μου ενταγμένο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον εισηγητή για αυτή την στιβαρή πραγματικά έκθεση. Σας ευχαριστώ. Σας παρακαλώ ε, τελευταίος ε, ομιλητής και λίγο σεβασμό και λίγη ησυχία στον ομιλητή παρακαλώ. Κυρία Νταντσίλα, κυρία Πρόεδρε, η Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της στρατηγικής της θέσης αλλά και λόγω των οικονομικών ε, ευκαιριών που προσφέρει και τη δυνατότητα για μια καλύτερη περιφερειακή ανάπτυξη που δίνει. Η στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα θα συνεισφέρει στη βελτίωση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της περιοχής, μια καλύτερη συνεργασία στην ε, έρευνα και στην εκπαίδευση, αλλά και για μια καλύτερη συνεργασία για την προστασία των φυσικών πόρων της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει τις χώρες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας για να δουν τι ενεργειακοί πόροι υπάρχουν, τι δυνατότητα υπάρχει για υφόρο ανάπτυξη και βελτίωση της περιοχής, της, της ζωής στην περιοχή και καλύτερη περιφερειακή ε, συνεργασία. Ε, ζητώ συγγνώμη από αυτούς που δεν πήραν τον λόγο στα πλαίσια της ΕΣ διαδικασίας Catch the Eye, αλλά δεν μπορούσα να τον πάρουν όλοι και τώρα τον λόγο έχει ο Επίτροπος Φίλε. Ευχαριστώ. να κάνω ε, Παρατηρήσει Το πρώτο το είπα και στην αρχή. Εκτιμούμε αυτή την επίκαιρη έκθεση για τη Μαύρη Θάλασσα. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσω αυτό το οποίο να καλωσορίσω αυτό το οποίο φάνηκε στη συζήτηση, τη σημασία που αποδίδουμε δηλαδή σε αυτή την περιοχή, τη σημασία που συμμερίζεται και η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τρίτον, αναμένω τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στρατηγική της Μαύρης Θάλασσας Λίγη ησυχία σας παρακαλώ λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Για να κλείσουμε τη συζήτηση δίνω το λόγο στον εισηγητή και σας ε, προτείνω να τον ακούσετε. Κυρία Πρόεδρε, είμαι πολύ τυχερός όχι γιατί ακούγομαι λόγω του θορύβου, αλλά γιατί με υποστήριξαν ουσιαστικά όλες ε, οι παρατάξεις όλες οι πολιτικές ομάδες. Όπως είπε στις πολύ εύστοχες παρατηρήσεις του και ο κύριος Μπροκ, η έκθεση την οποία θα ψηφίσουμε σε λίγο είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα διακομματικής πολιτικής συνεργασίας στο Κοινοβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πάσκολος ιδιαίτερος που απεδείχθη ιδιαίτερα δραστήριος και ενεργός θειασότης της πρότασης. Θα ήθελα να περιοριστώ σε αυτό το όνομα και να μην αναφέρω και άλλα γιατί θα ήταν άδικο για όσους τυχόν λησμονήσω. Σε ό,τι αφορά τη μοναδικότητα της περιοχής του Ευξηνού Πόντου, της ανάγκης να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διατυπώνουμε πολιτικές για την περιοχή αυτή. Πολύ σημαντικές ήταν και οι παρατηρήσεις βέβαια που αφορούσαν την αναγκαιότητα του έργου για τον των αεριού Ναμπούκο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον ε, Επίτροπο, τον ε, κύριο Φίλη, για τις παρατηρήσεις του και ιδιαίτερα γιατί αναφέρθηκε και στη θαλάσσια διάσταση. Μια πολιτική που διαμορφώνει του παρόντος Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει σίγουρα να υπάρξει και η διασύνδεση μεταξύ της, συνέργειας για, της στρατηγικής για τον Εύξηνο Πόντο και της στρατηγικής για το Δούναβ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ που ε, είσαστε ιδιαίτερα θαραλέως και προσπαθήσατε σε αυτή την οχλαγωγία μέσα, κύριε Σικτά, να μιλήσετε.